Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Αν δεν σας πειράζει, αρχίσουμε. Καλώς ορίσατε όλοι. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Ως πρώτος αντιπρόεδρος, έχω τη τιμή σήμερα να προεδεύω. Η πρόεδρος μας, κυρία Μακάβαν, κολλείται, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις αλλού και δυστυχώς με το πρωί Άρα, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση αυτής. Εφωνεί κανείς με την ημερήσια διάταξη. Όχι. Οπότε και εγκρίνεται. Δεύτερο θέμα. Σας θυμίζω αγαπητοί συνάδελφοι ότι στις 6 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο 8.30 με 10. Έχουμε κοινή συνεδρίαση έκτακτη τρεις επιτροπές, ε, ΔΕΒΕ, ε, ΑΦΕΤ και ε, ΔΓΟΑ για την παρουσίαση των πέντε υποψηφιωτήτων που λάβαμε για το βραβείο Σαχάροφ 2016. Ξέρετε ότι είναι το βραβείο που απονέμει το Κοινοβούλιο για την ελευθερία του πνεύματος. Τρίτο θέμα, στη μέση διάταξη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη. Le premier Πρώτο και μοναδικό ουσιαστικό θέμα στην σημερινή ημερήσια διάταξή μας είναι η ανταλλαγή απόψεων για ε, την αναθεώρηση ε, της συνένεσης αυτής με τον Επίτροπο κύριο Νέβεν Μίμητσα, τον οποίο έχω τη χαρά να καλωσορίζω Θυμίζω ότι το 2005 εγκρίθηκε η πρώτη Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη, η οποία για πρώτη φορά ορίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις κοινέ αξίες, αρχές, αλλά και τους στόχους της πολιτικής ανάπτυξης, όπου δεσμεύονται όχι μόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που υπογράφουν αλλά και τα κράτη-μέλη ε, ως πάροχοι της διμερούς ε, αναπτυξιακής βοήθειας. 11 χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 2015, και δεδομένου ότι έχουμε κοινέ προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή και οι μεταναστευτικές ροές, ε, αλλά και επειδή διαφέρουν οι χώρε αναπτυσσόμενε μεταξύ του, έχει έρθει η ώρα να αναθεωρηθεί αυτή η συνένεση και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και στι νέε πραγματικότητε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, ε, Άρχισε τον Ιούνιο μια δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση τη συνένεση αυτή, η οποία διαβούλευση ολοκληρώθηκε τέλη Αυγούστου. Επίση γνωρίζουμε ότι ήταν αυτό ένα από τα βασικά θέματα τη άτυπη συνεδρία των Υπουργών Αναπτυξιακή συνεργασία πριν από 15 μέρε, στην οποία παραβρέθηκαν και ο κύριο Μίμητσα όπω και η κυρία Μογκερίνη. Έχω λοιπόν τη μεγάλη χαρά και τιμή να δίνω το λόγο στον Επίτροπο κύριο Μίμητσα για να μοιραστεί μαζί μα τι πρώτε εντυπωσει που έχει ε, σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση, αλλά και να μας πει τι έγινε στην άτυπη Σύνοδο Υπουργών Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Επίσης, θα θέλαμε να μάθουμε λίγο περισσότερα για τις προετοιμασίες και πού βρίσκεται η ανακοίνωση που εκπονείται και θα καταθέσετε τέλη Νοεμβρίου. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. good Καλημέρα, κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, αγαπητοί συμμετέχοντες. Την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε ήταν τον Ιούνιο και είχα υποσχεθεί ότι θα ξανάρθω στην συνεδρίασή σας για να συζητήσω το μέλλον της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ακριβώς γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα υπήρχε μια κοινή αίσθηση ότι είναι και η ώρα η προθεσμία για την υλοποίηση των στόχων των αναπτυξιακών το 2030 ίσως. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε ήδη από τώρα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αντισώμενες ε, ε, ανισότητες, ε, μεταναστευτικές ροές αν προηγουμένου, ε, φτώχεια. Οι προκλήσεις της αναπτυξιακής ατζέντα χρειάζονται καλοσχεδιασμένες ευρείες λύσεις, αποφασιστική δράση, αμελητή. Τους επόμενους μήνες η δουλειά μας είναι ακριβώς αυτό να κάνουμε. Να παρουσιάσουμε δηλαδή μια αξιόπιστη και φιλόδοξη ευρωπαϊκή απόκριση στην ατζέντα του 2030 και να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε, να πάρουμε τα ενία, να δώσουμε το παράδειγμα σίγουρα πολύ σύντομα θα υπάρξουν ιδέες για την παγκόσμια αυτή στρατηγική και την εφαρμογή της και κατευθυντήριες γραμμές για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης από την ύπατη εκπρόσωπο που θα, καθοδηγήσουν, ε, θα μας καθοδηγήσουν στη νέα μας αυτή συνενετική πορεία. Παράλληλα, ε, υπό την αιγίδα του κ. Τίμερμαντς, μία ομάδα επιτρόπων δουλεύει για μια επικοινωνία για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον. Ούτω ώστε να δούμε πώ οι εσωτερικέ και εξωτερικέ πολιτικέ μα θα συνεισφέρουν στην εφαρμογή των ε, αναπτυξιακών στόχων. Επειδή, επειδή εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και εμείς στο εσωτερικό μας να προσπαθήσουμε για την πλήρη εφαρμογή των αναπτυξιακών στόχων, ειδικά σε ό,τι αφορά την ανισότητα, τη φτώχεια και την ε, άνηση ανάπτυξη. Το είπα και πριν. Σε ό,τι αφορά την βιωσιμότητα και την υλοποίηση και επίτευξη της βιωσιμότητας, είμαστε όλες αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, είμαστε στις τελευταίες φάσεις ε, προετοιμασίας των συστάσεών μας για μια αναθεωρημένη ευρωπαϊκή συνένεση για την ανάπτυξη και αυτό θα είναι στον πυρήνα των προσπαθειών μας για να εφαρμόσουμε τους στόχους ε, τους αναπτυξιακούς στις εξωτερικές μας δράσεις. Από την αρχή σκέφτηκα αυτή την ε, ανοιχτή και γενική διαδικασία θα ήθελα να τη δρομολογήσω. Καταρχάς ευχαριστώντας τα μέλη της Επιτροπής σας για την ε, συνεργασία και, την, ε, και το ζήλο και τη δέσμευσή σας. Αναπτύσσοντας τις ιδέες μας, κάναμε μια προσπάθεια να φτάσουμε και σε ένα ευρύτερο κοινό online, με σοβαρές συζητήσεις και στα πλαίσια τον Ιούνιο, της ημερίδας που έγινε στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο για την αναπτυξιακή, τα αναπτυξιακά θέματα και στο, στη Νέα Υόρκη σε ένα ευρύτερο φόρουμ και σύντομα θα δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα ε, καθώς και μία σύνοψη των 200 περίπου απαντήσεων που λάβαμε. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των απαντήσεων. Υπήρξε σαφή στήριξη για μια αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Συνένεση με βάση την ατζέντα του 2030. Αλλά η ανάγκη για μια αλλαγή με τις πορείας και ταχύτητα στις δραστηριότητε μας ε, προκύπτει ξεκάθαρα ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα γρήγορα και διαφορετικά. Αυτό προέκυψε και στις πρόσφατες συζητήσεις με τους επικεφαλείς ε, των διπλωματικών αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι τα αυτιά και τα μάτια μας στις χώρες εταίρους και στην άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Ανάπτυξης πριν από δύο εβδομάδες, στις 12 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Τέλος, μια νέα συνένεση για την ανάπτυξη βασίζεται στην ε, προσπάθεια την κοινή της Κομισιόν, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών επίσης. Και ελπίζω ότι αφού θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας, και την ε, ανακοίνωση στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα συμφωνήσουμε για μια νέα κοινή δήλωση ε, μαζί σας, δηλαδή εσείς και το Συμβούλιο. Ξέρω ότι στο εσωτερικό αυτής της Επιτροπής ετοιμάζεται ένα ψήφισμα μαζί με τους δύο συνεισηγητές που θα υιοθετήσει το Φεβρουάριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη σημερινή συζήτηση, ούτως ώστε να ενισχύσουμε αμοιβαία τη δουλειά που κάνουμε και στην ε, ανακοίνωση και στην έκθεση που ετοιμάζετε εσείς ιδίας πρωτοβουλίας. Είναι σημαντικό να έχουμε κοινέ απόψεις για τα βασικά θέματα. Σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε και το τι προτιθέμεθα να πετύχουμε και πώς ελπίζουμε να το υλοποιήσουμε αυτό. Πώς ελπίζουμε να το πετύχουμε, ας πούμε. Καταρχάς το πώς. Εμπνευστήκαμε από το προήμιο της ατζέντα του 2030 και την ανάγκη να συνδέσουμε τους ανθρώπους με την ευμερία, με τον πλανήτη και την ειρήνη. Είναι σαφές ότι οι καθολικές και παγκόσμιες αξίες που εγγράφονται στις ευρωπαϊκές συνθήκες και στο διεθνές δίκαιο, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα είναι οι θεμελιώδεις αρχές της ε, εξωτερικής μας δράσης ανά τον κόσμο. Οι βασικές μας δεσμεύσεις για να εξαλείψουμε τη φτώχεια σε όποια μορφή και αν υπάρχει και να μην αφήσουμε κανένα πίσω και εγκαταλελειμμένο, θα εξακολουθεί να εμπνέει όλες τις δράσεις μας θα συμφωνήσουμε, ελπίζω να συμφωνήσουμε, ότι η νέα συνένεση θα πρέπει να αντιμετωπίζει το θέμα αυτό της στόχιας, να την εξαλείψει. Σεβασμό στο περιβάλλον και κοινωνική βιωσιμότητα όλα μαζί. Όχι ως αντικρουόμενες προτεραιότητες, αλλά μέσα από συνέργειες. Επίσης, ε, θα πρέπει τα ωφέλη από τις δράσεις μας να μοιράζονται ε, πιο δίκαια ε, αντιμετωπίζοντας τις ανισότητες μεταξύ των χωρών και στο εσωτερικό των χωρών. Επίσης, θα πρέπει η πολιτική μας για την ανάπτυξη να είναι πολύ πιο συνεπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την, τον ηγετικό ρόλο που έχετε δείξει και παίξει σε αυτό το θέμα της συνοχής των πολιτικών ανάπτυξης. Και έχω καταγράψει ε, με μεγάλη προσοχή τα μηνύματα που προκύπτουν από το ψήφισμά σας τον Ιούνιο θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία σε βασικά θέματα όπως ε, το φύλλο, ιδεότητα, ε, ε, ενέργεια, επενδύσεις, μετανάστευση, κινητικότητα. Το να λειτουργήσουμε σωστά και να αντιμετωπίσουμε σωστά αυτά τα οριζόντια θέματα, θα, από αυτό θα εξαρτηθεί η επιτυχία και η επίπτωση που θα έχει η νέα συνένεση. Η εστίαση στις γυναίκες και στους νέους θα πρέπει να είναι μοχλή ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει απλώς να ωφελήσουν τις κατηγορίες αυτές. Και θα πρέπει να στο τονίσουμε πώς η ειρήνη και η ανθρωπιστική δράση ε, συμπληρώνουν και δεν έρχονται σε αντίθεση με τις αναπτυξιακές μας προσπάθειες. Η ατζέντα του 2030 μιλάει επίσης για τις εταιρικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα Επίσης συμφωνούμε ότι για να τα καταφέρουμε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η νέα συνένεση θα πρέπει να μας οδηγεί σε μια μετάβαση ε, προς μια πιο ε, αποτελεσματική κινητοποίηση όλων μας των πόρων. Η ατζέντα της Αντίσα Μπέμπα θα πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι σημαντική για την υλοποίηση την επιτυχή υλοποίηση των στόχων μας. Η αξία της βρίσκεται στην πληρότητά της, ε, στο, στο γεγονός ότι μιλάει για την βοήθεια, ανάπτυξη, κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων και ενίσχυση της διακυβέρνησης και κατάλληλων πλαισίων πολιτικής. Το να περάσουμε από τα δισεκατομμύρια στα τρισεκατομμύρια που χρειάζονται για να πετύχουμε αυτούς τους ευρύτατους αναπτυξιακούς στόχους ε, δεν θα γίνει εάν παραμείνουμε μόνο στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και στα όσα προβλέπει. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω με πολύ πιο έξυπνο τρόπο, χρησιμοποιώντας τμήμα τη, ούτως ώστε να μοχλεύσουμε και να ελκύσουμε και ιδιωτικές επενδύσεις ε, και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Από τότε που συναντηθήκαμε τελευταία φορά ε, υπάρχει πρόοδος σε αυτό. Ειδικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο, το ευρωπαϊκό ε, επενδυτικό σχέδιο για το εξωτερικό που εγγενίασε ο πρόεδρος Γιούνκερ πριν από δύο εβδομάδες ενώπιον του οίκου σας. Με αυτό το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ε, αυξήσουμε τις ξένες επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αντισώμενες χώρες, ιδίως στα ευπαθή κράτη όπου ο κίνδυνος είναι πιο μεγάλος και οι επενδυτές διστάζουν περισσότερο να πάνε. Το να λειτουργήσει αυτό το σχέδιο επιτόπου είναι μία από τις προσωπικές μου προτεραιότητες. Θα ξεκινήσουμε με την Αφρική και την Ευρωπαϊκή Γειτονία και θα βασιστούμε στα υπάρχοντα εργαλεία, τα οποία όμως βελτιώνται συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε με 3,4 δις από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και ελπίζουμε να ελκύσουμε μέχρι 44 ε, δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις. Αλλά χρειαζόμαστε βεβαίως και τα κράτη-μέλη και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βάλουν και αυτά τον οβολό τους. Και χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας. Αν τα κράτη-μέλη και οι υπόλοιποι εταίροι σεβαστούν τι δεσμεύσεις, το συνολικό ποσό των επενδύσεων μπορεί να φτάσει και τα 88 δισεκατομμύρια. Χρειαζόμαστε μία πιο συντονισμένη προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινή δράση, κοινό προγραμματισμό, πολύ πιο έντονο μάλιστα. Πολλά άλλαξαν από την υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Συνένεσης του 2005. Όχι μόνο προέκυψε η Σύνθηκη της Λισαβόνας, αλλά και διάφορες παγκόσμιες προκλήσεις που, αποτελούν, που είναι τεράστιο θέμα και απαιτούν συλλογική απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το συντηρητικό πλεονέκτημα που έχουμε και, την, και να αντλήσουμε δύναμη από την ποικιλομορφία μας. Οι εταιρικέ σχέσεις ε, σημαίνει διαφοροποιημένες εταιρικέ σχέσεις με διαφορετικές χώρες που βρίσκονται σε διαφορετική φάση ανάπτυξης. Μαζί με την ανακοίνωση για την αναθεωρημένη συνένεση θα παρουσιάσουμε και τις προτάσεις ε, για τις μελλοντικές μας σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ. Μετά την ε, εκπνοή της Συμφωνίας Κοτονού. Οι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε και οι εύθραυστε χώρε θα πρέπει να είναι στο κέντρο των αναπτυξιακών μα προσπαθειών. Ε, πρέπει να συγκεντρωθεί κυρίω εκεί η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Παράλληλα, οι χώρε μεσαίου εισοδήματο θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο για να εφαρμόσουν του στόχου του αναπτυξιακού, μέσω όμως διαφορετικών μορφών συνεργασίας, ε, εμπόριο, άμεσες ξένες επενδύσεις, τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη για πολιτική με σκοπό να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, υπό τη νέα Ευρωπαϊκή Συνένεση θα πρέπει να ξεπεράσουμε ε, την απλή μέτρηση των αποτελεσμάτων της βοήθειας. Θα πρέπει να περάσουμε στη διαφάνεια, ε, στο follow-up, στην αναθεώρηση και οι δαπάνε για την ανάπτυξη θα πρέπει να ε, γίνονται με το πιο, το πιο αποτελεσματικό τρόπο και να προσαρμόσουμε τα εργαλεία και τους μεθόδους, τις μεθόδους εργασίας. Θα πρέπει εμείς να είμαστε πρωταθλητές ε, διαφάνειας μέσω ενός κοινού πλαισίου για την ανάπτυξη ε, και να υποστηρίξουμε, υποστηρίξουμε τους εταίρους μας για να συνδέσουν τους πόρους για την ανάπτυξη με τα αποτελέσματα υποστηρίζοντας το δικό του στατιστικό δυναμικό. Εν συντομία, Αυτές είναι οι θεμελιακές αρχές που στηρίζουν το σχέδιο πρότασής μας. Περιμένω να ακούσω αν συμφωνείτε με αυτά που σας παρουσίασα, το πώς και το τι. Και να μου πείτε αν έχω συμπεριλάβει όλα τα βασικά στοιχεία. Ε, στηρίζομαι στην ειλικρή, ειλικρινή ε, συνεισφορά σας ούτω ώστε να δημιουργήσουμε την καλύτερη βάση για μια νέα ευρωπαϊκή συνένεση. Μια συνένεση που θα λαμβάνει υπόψη την περιπλοκότητα της ατζέντα του 2030, που βασίζεται στο θρύλο ε, που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ηγετικέ της προσπάθειες στον χρόνο της ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ και περιμένω με ανυπομονησία να ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, ανοίγει τώρα η συζήτηση. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους δύο συνεισηγητές μας, τον Μπόγκταν και τον κύριο Νόισερ. και μετά οι σκιώδες συγητές. Ο Μπόγκταν Βέντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, η αναθεώρηση του κοινού οράματο της Ευρωπαϊκής ένωση τη αναπτυξιακής πολιτικής μέχρι το 2030 είναι μείζον ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της. Προσωπικά είμαι πεπισμένο ότι έρχεται την κατάλληλη στιγμή από τη μια η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές και από την άλλη αλλάζει ε, και το πλαίσιο των προτάσεων. Η αναθεώρηση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Συνένωσης για την Ανάπτυξη είναι μία από τις πολιτικές που καλούμεθα να ξαναδούμε. Έχουμε αναθεωρήσει το παλιό ε, κείμενο και έχει αρχίσει η εκπόνηση του νέου κειμένου και θα ενταχθούν και συνολικοί στόχοι για την ανάπτυξη ενόψη του 2030. Θα ήθελα να σας ρωτήσω μερικά πράγματα. Το πρώτο αφορά τη σύνδεση της Ευρωπαϊκής Συνένεσης με την ανάπτυξη και την αναπτυξιακή βοήθεια. Δεν θα πρέπει να έχετε κάποιες κοινέ αναφορές για να συνδεθεί καλύτερα η ανθρωπιστική βοήθεια με την αναπτυξιακή βοήθεια. Επόμενη ερώτηση. Αφορά τον κοινό προγραμματισμό της ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Μέχρι τώρα εφαρμόζεται αυτή σε 55 αναπτυσσόμενες χώρες. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν ε, κατά τη γνώμη σας για να ενισχυθεί ε, και να ενθαρρυνθεί αυτή η πρακτική και πώς θα βρίσκεται ανάκλαση στη νέα συνένεση. Και τελευταία σχόλια, πώς συνδέεται η μετανάστευση με την ανάπτυξη και πώς μπορεί να ενισχυθεί σε πρακτικό επίπεδο αυτή η σύνδεση. Δηλαδή, θα πρέπει εμείς να καταπολεμήσουμε τις αιτίες της μετανάστευσης που είναι η φτώχεια, η αστάθεια, η πόλεμη, η διαφθορά, η ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε Βέντα. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Νόρμπερτ Νόης. Ja, vielen Dank, äh, Herr Kommissar. στο λόγο τώρα στους και ηγητές, αν επιθυμούν. Ο Σνάφος Γκέρενς πρώτος. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε σήμερα για τη συνένεση ε, και έχουμε να κάνουμε και με θέματα μεθόδου και με θέματα ουσίας. Για την ουσία θα επιθυμούσα το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και και ΜΚΟ να συμφωνήσουν για τον ίδιο ε, ορισμό του τι εστί ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν όλοι έχουμε την ίδια αντίληψη ε, για την ανάπτυξη. Για μας εδώ στο Κοινοβούλιο Πρόκειται κατά κύριο λόγο για την καταπολέμηση της στόχιας με εταιρικό πνεύμα, με εταιρική σχέση και θέλουμε να δούμε τους εταίρους μας να χειραφετούνται και κάποια στιγμή να μην έχουν ανάγκη και να μην εξαρτώνται από τη βοήθειά μας. Βλέποντας όμως τις διάφορες αντιδράσεις, κάθε φορά που βλέπουμε μια καταστροφή, μια κρίση προσφύγων, λέμε, α ναι, να κάνουμε κάτι παραπάνω για την ανάπτυξη. Έμας ε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το τονίζουμε αυτό και να το απαιτούμε. Και όταν δεν υπάρχουν θεομηνίες και καταστροφές γνωρίζουμε πλήρη αδιαφορία. Δεν καίγεται καρφή σε κανένα. Θα πρέπει λίγο λοιπόν να δώσουμε περισσότερη δύναμη και ισχύ σε εκείνους που συνεχώς επιμένουν και επαναλαμβάνουν ότι θα πρέπει να επιτεθούμε στη ρίζα του κακού. Η φτώχεια προφανώς προκαλεί σειράξεις οι σειράξεις προκαλούν ανθρωπιστικές κρίσεις και η ανθρωπιστική δράση είναι απάντηση σε όλες αυτές τις αποτυχίες. Τώρα εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα της έλλειψης, ανάληψης ευθυνών απέναντι σε αυτά τα μεγάλα θέματα και φαινόμενα. Δεν φταίτε εσείς, ούτε η γενική σας διεύθυνση, ο γενικός διευθυντής, οι ε, υπηρεσίες, το κοινοβούλιο, αλλά η σύνολη διεθνής κοινότητα και σίγουρα κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέκαθεν υποτιμούσαν τη σημασία της αναπτυξιακής πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε, πιστεύω, σε ένα κοινό ορισμό στο τι πρέπει να κάνουμε κατά πρώτο λόγο και να καταρτήσουμε και ένα κατάλογο των μέτρων που ακολουθούμε στην πολιτική ανάπτυξη που ε, το πολύ πολύ τα συμπτώματα θεραπεύουν, όχι την αιτία. Και είναι και επενιχρή πόρη τώρα και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε και τις αφρικανικές κυρίως χώρες και ιδιαίτερα όλες αυτές τις χώρες που είναι στην άμεση σφαίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατρανώνονται διάφορες προθέσεις αύξησης ε, της συνεισφοράς, αλλά όταν έρχεται η ώρα να τα μετρήσουμε τα χρήματα δεν βγαίνουν. Και τίθεται και ένα θέμα ε, αξιοπιστίας. Και πάντα εξαγγέλνουμε διάφορα ωραία πράγματα που ποτέ δεν επαληθεύονται και δεν υλοποιούνται. Από πλευρά μεθόδου λοιπόν θα πρέπει να είμαστε από τη μια αυστηροί ε, ω προ τον ορισμό αλλά και ω προ τι δεσμεύσει που αναλαμβάνουμε. Σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής μας σχεδόν επαναλαμβάνω αυτό το πράγμα και θα συνεχίσω να το επαναλαμβάνω ε, εφόσον δεν λύνεται το πρόβλημα. Πώς θα το λύσουμε. Να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι και αλλιώς, γρήγορα θα συμφωνήσουμε και μεταξύ μας και να καλέσουμε και τα κράτη-μέλη και τις ΜΚΟ. Να δούμε ποια θα μπορούσε να είναι η βάση μεγαλύτερης αξιοπιστίας πολιτικής αυτής. θα συμφωνήσουμε για κάποιες αρχές. Όλες αυτές οι κοινοτυπίες και τα κούφια λόγια που ακούμε και τις μεγάλες διασκέψεις, ε, τα SDG, ωραία. Ε, τι είναι η βιώσιμη στόχη, η αναπτυξιακή, το είπατε κι εσείς. Είμαστε όλοι αναπτυσσόμενες χώρες, το έχουμε καταλάβει ε, για την αηφορία και τη βιωσιμότητα. Το έχουν καταλάβει και τα 28 κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χαράξει καμιά στρατηγική αντίστοιχη, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν όλοι και να στοιχηθούν και 28 πίσω από μια κοινή γραμμή. Αν έχουμε λοιπόν κοινή ανάγνωση, αν θέλουμε να έχουμε τέτοια ανάγνωση, διαπιστώνουμε ότι όλες οι χώρες του κόσμου υπόκειται στην παγκοσμιοποίηση που έχει διπλή επίπτωση από τη μια μειώνει τις διαφορές ανάμεσα στις χώρες, αλλά εντείνει και αυξάνει τις διαφορές στο εσωτερικό ε, μιας χώρας. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Θα πρέπει ε, τα τρία θεσμικά όργανα και να συμφωνήσουν για να καταλάβουν ότι η μέθοδος που ακολουθούμε μέχρι τώρα είναι ξεπερασμένη. Δεν προσφέρεται για να αντιμετωπίζει τα σημαίνα προβλήματα. Σας λέω λοιπόν ειλικρινά, εάν δεν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για αυτές τις βασικές αρχές τις λίγες και δράσεις βασικής, πολύ αμφιβάλλω ότι θα έχουμε αξιόπιστο αποτέλεσμα στην αναθεώρηση της συνένεσης αυτής και θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο κρίμα. Επανειλημμένα έχω πει και το ξαναλέω και το ξαναζητώ. Και δεν μιλώ μόνο εξ ονόματος της ομάδας μου, των φιλελευθέρων, αλλά όλοι συμμεριζόμαστε αυτή την ανησυχία. Τι θα κάνουμε τελικώς έτσι ώστε αυτές οι πανηγυρικές διακηρύξεις και δεσμεύσεις ε, να τηρηθούν. Έχουμε κανένα μέσο παρακολούθησης ελέγχου. Να δούμε τι γίνεται ας πούμε σε επίπεδο ευρωπαϊκού εξαμήνου. Αυτή αυξάνονται τα ελλείμματα των κρατών να προσκαλούνται στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να λογοδοτούν. Αφού όλοι θέλουμε να συγκλίνουμε προς την ίδια πολιτική, η πολιτική ανάπτυξης είναι λιγότερο σημαντική ή καθόλου. Αν είναι σημαντική θα πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα κοινά εργαλεία για να τα ελέγχουμε. Που αυτά ήδη φαίνεται ότι αποδίδουν αλλού. Ζητώ λοιπόν στην πολιτική αυτή να υιοθετήσουμε μια τέτοια προσέγγιση που να την δέχονται όλοι αλλά να δεσμεύονται όλοι και να ισχύουν τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης προς όλους. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για να πιστεύουμε ότι η νέα συνένεση μπορεί να επιτύχει καμιά αλλαγή. Ε, πραγματικά εδώ διακυβεύεται η αξιοπιστία μας. Από τη μια εμείς εδώ ε, υπερασπιζόμαστε μια πολιτική, όλα αυτά που λέμε δεν ενδιαφέρουν κανέναν, καρφί δεν καίγεται στο Συμβούλιο, διότι κάποιες χώρες, όχι όλες, εντάξει, αδιαφορούν. Ε, τι άλλαξε από το 2005, Σα είπα, ποιες είναι οι σταθερές σταθερά είναι ότι δεν τηρούμε τι υποσχέσει μα. Πρέπει να τερματεί αυτό. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι η παγκοσμιοποίηση πραγματικά έχει εδρεωθεί και κυριαρχεί παντού σε όλε τις πολιτικές. Παντού. Έχει αντίκτυπο μέχρι και στην ιδιωτική ζωή του καθενό μα. Αυτό που άλλαξε επίση είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι αιστείε κρίση και ανάφλεξη. Και αποτέλεσμα αυτό τη αδυναμίας πρόληψη των σειράξεων γέρου. Άλλο που άλλαξε, οι ανισότητες αυξάνουν. Θα πρέπει να ε, αδράξουμε όλα τα μέσα που έχουμε, να τηρούμε τις υποσχέσεις μας και τις δεσμεύσεις μας, παρά να πολλαπλασιάζουμε τις αποτυχίες. Για το λόγο αυτό επίσης ζητώ να συμμετέχουν περισσότερο οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις στη διαδικασία αυτή, που θα πρέπει να είναι η συνείδηση όλης αυτής της πολιτική Και με τέσσερι εταίρους ισχυρού, Συμβούλιο, Κομισιόν, εμείς και ΜΚΟ, θα τα καταφέρουμε. Ήθελα να τα πω αυτά, ε, να συμφωνήσουμε επί της ουσίας, επί της μέθοδου. Και αν αυτό γίνει τελικά μια φάρσα και ε, ένα γελίο πράγμα, να μην συμμετέχει πια το Κοινοβούλιο. Η κυρία Θεοχάρους έχει το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Chair.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 Ευχαριστώ κύριε Θεοχάρους. Μαρία Όλμπους. Μαρία Χοέμπουχα από τους Πρέσινους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τα όσα μας εκθέσατε εδώ. Είπατε ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και να μην ξεχνάμε το περιβάλλον, το κλίμα και να μην αφήνουμε κανέναν αβοήθητο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και εγώ ήμουν μέλος αντιπροσωπείας που ακούσαμε προηγουμένως και βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που είναι αβοήθητοι και πρέπει να τους βοηθήσουμε. Άρα από πλευρά στόχων ε, βιώσιμοι ε, στόχοι θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Τους χαρακτήρισε πραγματική επανάσταση ο Σάρλ Γκέρενς και είναι τέτοια αν καταφέρουμε να του εφαρμόσουμε με μέθοδο. Και για την αναπτυξιακή συνεργασία θα ήταν ενίσχυση τη εικόνα τους ε, έναντι άλλων τομέων εξωτερικής πολιτικής και ένα ισχυρό μήνυμα ότι η αναπτυξιακή συνεργασία δεν θα πρέπει να ε, είναι κάτι που αντιλαμβανόμαστε από πλευράς ασφάλειας και μόνος, αλλά είναι ε, μια βάση η στόχη αυτή βιώσιμη και για το περιβάλλον και για το εμπόριο και για τη δράση μας. Θα πρέπει να δούμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να έχουμε ε, δίκαιη και αποτελεσματική συνδιαχείριση ε, των παγκοσμίων ε, δημοσίων αγαθών. Τι σημαίνει αυτό για μένα. Ότι η αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να ενταθεί, πρέπει να αυξηθεί και η ανανεώση αυτής της συνένεσης αποτελεί ευκαιρία για μας αλλάξουμε τη χορογραφία της συνεργασίας των κρατών μας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπως είπε ο Σαλγκέρενς να βρούμε νέες μεθόδους να εφαρμόσουμε. Διότι αν δούμε πώς έχει σήμερα η κατάσταση, ε, πιστεύω και εγώ ότι να βρουμε νεες μεθοδους να εφαρμοσουμε διοτι αν δουμε πως εχει σημερα η κατασταση πιστευω και εγω οτι δεν μπορουμε να συνεχισουμε με τις ίδιες μεθόδους που έχουμε ακολουθήσει ως τώρα. Ε, πολύ σύντομα να σας αναφέρω μερικά σημαντικά θέματα μια συνεκτική πολιτική, ουσιαστική, συνενοημένη αναπτυξιακή βοήθεια, αντί ο καθένας κοντόφθαλμα και ε, βράχει πρόθεσμα να εξυπηρετάει οι ίδια συμφέροντα. Η αναπτυξιακή και εμπορική πολιτική είναι σημαντική για την παγκόσμια ανάπτυξη και βεβαίως ε, δεν θα πρέπει να λείπει από τη συνένεση. Η πολιτική ασφαλεία επίσης. Έχω πάντα την αίσθηση, πρέπει να πω, ότι τα ευρωπαϊκά ίδια συμφέροντα κυριαρχούν ε, πέραν του πρωταρχικού στόχου της αναπτυξιακής βοήθειας και δεν θα πρέπει να είναι αυτός ο σκοπός. Ε, οφείλω βέβαια να αναγνωρίσω ότι στην ασφάλεια θα πρέπει να ενδαθούν οι προσπάθειές μας, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι από τα λεφτά που έχουμε στη διάθεσή μας για την καταπολέμηση της φτώχειας. Δεν νομίζω. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ένδυα, πρέπει να αυξηθεί η ε, χρηματοδότηση. Αλλιώ δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ ούτε να ελεγχθεί το φαινόμενο και το πρόβλημα τη ασφάλεια. Εκεί θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε πάρα πολύ προσεκτικά από ποια κονδύλια παίρνουμε χρήματα για να τα δίνουμε στην πολιτική ασφαλείας. Δεν θα πρέπει να πληρώσει τα σπασμένα ή καταπολέμηση τη φτώχεια. Αναπτυξιακή συνεργασία λοιπόν κατά την άποψή μου δεν είναι ένα εργαλείο για να ασκούμε μεταναστευτική πολιτική. Είναι ξεχωριστό κεφάλαιο. Η υλοποίηση της ατζέντας του θεματολογίου 2030. Εγώ εδώ είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την καταπολέμηση της φτώχειας. Είπατε ότι δεν μπορεί να είναι μοναδική μας ενασχόληση ή ερμοδιότητα, αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά που έχουμε κρίση να λέμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια. Ενώ έχουμε στόχο από τον οποίο έχουμε ρίσει όλοι, το 0,7% του ΑΕΠ να πηγαίνει στην αναπτυξιακή βοήθεια που δεν τον έχουμε πετύχει. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα χρόνο διάγραμμα για να τηρηθεί και αυτός ο στόχος του 0,7%. Επίσης, θα πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα τη φορολόγηση ε, στις χώρες αυτές με τις οποίες συνεργαζόμαστε και να μην υπομονωμεύονται από κάποιες εμπορικές συμφωνίες όλα αυτά. Όταν ζητάμε ας πούμε, ε, πρόσβαση στις αγορές με κατάργηση των εισαγωγικών δασμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δίνει και το καλό παράδειγμα στην καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Ε, διαφάνεια ακούστηκε προηγουμένως είναι κάτι το οποίο ε, δεν θα πρέπει να λείπει από τη συνένεση. Έρχομαι τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας είναι πάντα ο συνομιλητής μας όταν λέμε ότι δεν μας φτάνουν τα κονδύλια, τα αναπτυξιακά της επίσημης βοήθειας κρατικής, χρειαζόμαστε ιδιώτες. Βεβαίως μπορούν να βοηθήσουν επενδυτές εκεί, αλλά θα πρέπει να ξεφύγουμε από την ιδέα ότι μια επένδυση θα πρέπει να ε, σημαίνει και ε, ωφέλεια για το λαό της χώρας. Θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι συνθήκες επένδυσης για να εγγυηθούμε τη βοήθεια και την ωφέλεια για τους κατοίκους αυτών των χωρών. Όλων. Και όλους είπατε να μην αφήσουμε κανένα στην άκρη. Ωραία δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε ακόμα για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Θα πρέπει να δούμε αν πιάνουν τόπο τα χρήματα και αυτό γίνεται και με κανόνες δεσμευτικούς και σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς και οικολογικούς κινδύνους που πρέπει να ε, περιορίζονται. Άρα αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να δείξουμε ε, θάρρος για να αλλάξουμε νοοτροπία και σκέψη και συνδέεται αυτό και με τη συζήτηση για με, την εποχή μετά το Κοτονού, τις νέες σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών ΑΚΕ κτλ. Εκεί χρειάζονται θαραλέα βήματα και έτσι θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε και με αισιοδοξία στο μέλλον. Θάρρος χρειάζεται, αλλιώ θα αφήσουμε και κάποιους στην άκρη και δεν θα καταφέρουμε να τους συμπεριλάβουμε όλους και αυτοί θα είναι τα μελλοντικά προβλήματα ή θα δημιουργήσουν τα προβλήματα του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Merci, cher. Ευχαριστώ, Έχουμε τρεις ακόμη ομιλητές. Θα τους ακούσουμε και εν συνεχεία ο Επίτροπος θα μας απαντήσει. Ο κύριος Λίτς. Καλημέρα, Επίτροπε, και ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας και για το πνεύμα των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων που παρουσιάσατε στο ΝΟΙΕ. μαζί με τον Τίμερμαν, σε εσά, την κυρία Μοντερίνη, ε, έχουμε παρακολουθήσει το πώς εξελίσσονται αυτοί οι στόχοι. Όπως είπατε και εσείς, η κατάσταση αυτή ε, είναι μια κατάσταση ρευστή εν εξελίξη, Όλοι μαζί θα πρέπει να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους και τώρα θα πρέπει να το καταφέρουμε μέσω πραγματικής δράσης. Γι' αυτό μου άρεσε αυτό που είπατε, το να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, να έχουμε μια συνεπή προσέγγιση, να επικεντρωθούμε στις γυναίκες ε, και το κάντε την ε, αναπτυξιακή χρονιά και να συντονίσουμε τις αναπτυξιακές προσπάθειες με τα κράτη-μέλη. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο πράγματα σε κάτι που είπε ο κύριος Γκέρενς καταρχάς. Τα κράτη-μέλη, το έχουμε πει πολλές φορές, πώς θα χρηματοδοτήσουμε την αναπτυξιακή μας βοήθεια, από πού. Το 0,7 είναι ακόμα επίκαιρο. Το πληρώνει μόνο Ηνωμένη, το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο μάλιστα φεύγει όπου να είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται με αυτό το 0,7 αναπτυξιακής βοήθειας. Έχουμε σημάδια από άλλους επιτρόπους και από τον προλογισμό ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα υλοποιήσουμε αυτό το στόχο του 0,7%. Και κάτι πρακτικό. Έχουν γίνει πολλές μεγάλες διασκέψεις για το θέμα της ανάπτυξης. Κάναμε συζητήσεις για το θέμα των κλωστοφεντουργικών και των ρούχων. Ε, διάφοροι φοιτητέ ε, τις ημέρες ανάπτυξης ε, έθεσαν το θέμα. Αν πρέπει να πληρώσουμε έστω και ένα ευρώ παραπάνω προκειμένου να αγοράσουμε ρούχα τα οποία δεν τα φτιάχνουν παιδιά. Από ό,τι κατάλαβα, τα κράτη-μέλη προσπαθούν να αναλάβουν δράση. Ε, η Γερμανία, ε, Σουηδία, Δανία, κατοχώρες θέλουν μια κοινή προσέγγιση, θέλουν να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από ό,τι άκουσα από τα κράτη-μέλη, γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Εσείς πώς το βλέπετε. Επίση κάναμε μια μεγάλη και πολύ ωραία διάσκεψη μαζί με την Κομισιόν για την έκθεση για τι κυβερνητικέ πρωτοβουλίε. Ε, έγινε πολύ έντονη προσπάθεια από την Κομισιόν. Η έκθεση αυτή θα δημοσιευθεί, άραγε θα την πάρει κανένα στα σοβαρά. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς βλέπει την ανάπτυξη από τη μία, το εμπόριο από την άλλη. Πιστεύετε ότι είναι καλό να, συνεργαστούμε, ή συνεργαστείτε με άλλους επιτρόπους για να προωθήσουμε τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να προχωρήσετε για να πετύχουμε αυτού του στόχου και για τα κράτη-μέλη αλλά και για του πληθυσμού των χωρών αυτών. Για τα χρηματοδοτικά μέσα. Να πω σε κάτι, να πω σε κάτι τεχνικό αλλά σημαντικό. Ε, το συζητήσαμε και στην ομάδα μα. για τα χρηματοδοτικά μέσα για την ασφάλεια. Στι 5 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μία πρόταση για να τροποποιήσει το εργαλείο ε, συνεισφορά στην σταθερότητα και ειρήνη, ε, κοινή ανακοίνωση ούτω ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να προλάβουμε τις κρίσεις. Ε, ε προβλέπουμε χρήματα για εξαιρετικές περιπτώσεις για να δώσουμε σε χώρες ε, εταίρους. Δύο ερωτήσεις έχω. Γιατί η Κομισιόν υιοθέτησε έναν αρνητικό κατάλογο και όχι θετικό κατάλογο για να καθορίσουμε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις. Δεν θα ήταν εύκολο, πιο εύκολο να βρούμε αυτά τα κονδύλια και να τα διαιρέσουμε ανάλογα με τις δράσεις. Η Κομισιόν ε, κάνει μια πρόταση που βασίζεται σε μια διπλή νομική βάση. Άρθρα 209.1 και 212.2 που είναι η νομική βάση για την αναπτυξιακή συνεργασία. Γιατί η Κομισιόν θέλει το χρησιμοποιήσει αυτά τα άρθρα 209 και 212 αντί για τα άρθρα 30 και 31 που είναι η νομική βάση για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Δεν θα είχε περισσότερο νόημα για τους στόχους της πρότασης να χρησιμοποιήσει το 30 και το 31. Ε, δηλαδή να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίζει στρατιωτικούς φορείς. Και εδώ συνδέεται με αυτό που είπατε για την ε, παγκόσμια στρατηγική της Μογκερίνη. Πώς συνδέεται αυτή η στρατηγική με το κλίμα. Το κλίμα νομίζω επισκιάστηκε λιγάκι ε, ω θέμα. Αλλά νομίζω ότι το κλίμα είναι και μια, μας είναι και μια θαυμάσια ευκαιρία για ανάπτυξη. Ε, δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε την ε, επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια μέσω του κλιματικού πακέτου που συμφωνήσαμε στο Παρίσι. Ευχαριστώ. Ε, επόμενος συνάδελφος, ο κ. Γκερέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στην αρχή της παρέμβασής σας μας είπατε ότι είμαστε, εν πλήρη, είμαστε σε φάση πτήσης, ας πούμε, σε διαβούλευση, σε διάλογο, με διάφορους συνομιλητές, κοινωνικούς, θεσμικούς, για τη μελλοντική αναθεώρηση αυτής της περίφημης συνένεσης. Μας είπατε ότι υπάρχει μια μεγάλη αποδοχή της ανάγκης για να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Από τη μία γίνεται μια θετική αξιολόγηση για το πόσο λειτουργήσε μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Συνένεση υπό την έννοια ότι επέτρεψε να συντονίσουμε τη δράση των διαφόρων φορέων θεσμικών και κοινωνικών. Και από την άλλη σημειώσατε τις αλλαγές που έγιναν σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι αλλαγές που έγιναν στους κοινωνικούς αυτούς εταίρους και όλα αυτά απαιτούν αυτή την αναθεώρηση. Γι' αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατ' επανάληψη μίλησε για την ανάγκη να γίνει αυτή η αναθεώρηση και χρησιμοποιείται πάντα αυτός ο όρος αναθεώρηση για να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται για να δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική συνένεση από την αρχή, αλλά να κρατήσουμε αυτό που λειτουργήσε παλιά, ε, καλά μέχρι τώρα από τη συνένεση και να βάλουμε τις αλλαγές που είναι απαραίτητες ούτως ώστε να δώσουμε μια νέα όθηση σε αυτή την ε, αναπτυξιακή συνεργασία σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο σήμερα από ότι το 2005. Τώρα για τους λόγους ε, αναθεώρησης. Ο ίδιος ο Επίτροπος μίλησε για διάφορους λόγους. Συμφωνώ και συμφωνούμε γενικά όλοι μας με αυτό. Ο κύριος Γκέρες μας είπε ο, ένα βασικό θέμα για την έννοια της ανάπτυξης. Ότι όλοι σε κάποιο βαθμό είμαστε αναπτυσσόμενες χώρες με διαφορετικές ανάγκες και με διαφορετικές στρατηγικές και με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. Όμως, άλλαξε η έννοια υπό την, υπό τη λογική ότι παλιότερα θεωρούσαμε ότι υπήρχαν χώρες οι οποίες χρειαζόταν αναπτυξιακή βοήθεια και χώρες οι οποίες έδιναν την αναπτυξιακή βοήθεια και ήταν δύο διαφορετικοί κόσμοι που κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες. Αντίθετα, ο κόσμος τώρα είναι πολύ πιο περίπλοκος, πολύ πιο σύνθετος. Υπάρχουν όμως και καθαρά ευρωπαϊκοί λόγοι γι' αυτό. Η εμφάνιση μιας παγκόσμιας στρατηγικής που θα την παρουσιάσει η ύπατη εκπρόσωπος τα διάφορα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν από το λεγόμενο Migration Compact, από το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, όλα αυτά συνδέονται με την πολιτική μας, την εξωτερική πολιτική, εν το συνόλο της. Και ό,τι σημαίνει αυτή η πολιτική για την αναπτυξιακή συνεργασία. Για μένα τώρα, για αυτά που με μένα με απασχολούν, επειδή είμαι και εισηγητής για την ανθρωπιστική βοήθεια, θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο ε, Ανέφερε και ο κύριο Γκέρες και άλλοι συνάδελφοι ότι ο δεσμός ανάμεσα στην αναπτυξιακή δράση και βοήθεια και την ανάπτυξη είναι ένας δεσμός τελείως διαφορετικός από αυτόν που υπήρχε παλιότερα πριν χρόνια. Οι ανθρωπιστικέ κρίσει είναι όλο και περισσότερο κρίσεις που είναι μεγάλης διάρκειας όλο και περισσότερο είναι κρίσει που προέρχονται από συγκρούσει, σειράξει, πολέμους κτλ. Και οτιδήποτε είναι αναπτυξιακή συνεργασία που έχει σαν σκοπό την πρόληψη των σειράξεων και την επίλυση των σειράξεων και οτιδήποτε είναι αναπτυξιακή συνεργασία για την έξοδο από αυτές τις ανθρωπιστικές κρίσεις, αυτός ο δεσμός θα πρέπει να ενισχυθεί, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε, θα πρέπει να του, να του εμφυσίσουμε μια νέα πνοή. Φυσικά, εγώ αυτά τα λέω εγώ τώρα, ε, γιατί είμαι εισηγητή, αλλά φυσικά δεν τα έχω πει μόνο εγώ, τα έχουν πει και άλλοι πριν από μένα. Θέλω όμως να το τονίσω έστω και τώρα ε, αυτό το θέμα και θέλω να μιλήσω και για την πρόληψη και για την ανθεκτικότητα. Και η πρόληψη των φυσικών καταστροφών, όπως και η πρόληψη των σειράξεων, και η επίλυση των σειράξεων συνδέεται με την οικονομική και θεσμική ενδυνάμωση. Ε, είναι σημαντικό για να επιλύσουμε τις παρατεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις. Και όλα αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στην αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Συνένεση. Όλα αυτά ενδιαφέρουν πάρα πολύ και το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μας και εμένα τον ίδιο προσωπικά πρέπει να υπάρξει αυτή η ενίσχυση αυτού του δεσμού για τον οποίο σας μίλησα. Ευχαριστώ αγαπητή συναδελφέ. Η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε σήμερα να μοιραστείτε τις απόψεις σας μαζί μας. Ακούγοντας τούτη τη συζήτηση, νομίζω μπορούμε να συμπεράνουμε και μπορώ να το πω και εγώ στη τελευταία μάλλον ομιλήτρια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγάλες προσδοκίες και επιθυμεί να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να βοηθήσουμε πραγματικά να καταπολεμηθεί η φτώχεια και να αντιμετωπίσουμε και άλλες προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή ε, στο νέο παγκόσμιο πλαίσιο για το 2030. Υπάρχει ένας κίνδυνος στον οποίο αναφέρθηκαν πολλοί ομιλητέ. Είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ πάρα πολύ. Ότι δηλαδή τώρα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πέφτουν όμοιροι άλλων πολιτικών ή αναπτυξιακές πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικαλείται ένα ηγετικό ρόλο στην αναπτυξιακή βοήθεια και πώς θα το διατηρήσει όταν βλέπουμε να ξυλώνεται μέσω το μέσο εργαλείο το εργαλείο ε, και αποψηλώνονται ε, αυτά τα μέσα που έχουμε για την καταπολέμηση της φτώχειας και για την αναπτυξιακή βοήθεια. Και είναι και τεράστιες πέρα από τη φτώχεια, κλιματικέ αλλαγές, η διάβρωση ε, των παγκοσμίων δημοσίων αγαθών. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σχέση με την έννοια της ε, συνεκτικότητας και συνέπειας των πολιτικών για την ανάπτυξη. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολιτικές ε, σε άλλους τομείς που βοηθούν την ανάπτυξη, ε, αλλά τώρα βλέπουμε να παίρνει ένα χαρακτήρα ε, στραμμένο περισσότερο προς την ασφάλεια αναπτυξιακή συνεργασία. Δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Και κάθε πρώτη Ευρωπαϊκής ε στρέφεται προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε όλο και λιγότερο χώρο και χρήμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και μάλιστα της ρίζες και τα αίτια του κακού. Εσείς ως αρμόδιος επίτροπος θα πρέπει να δείξετε μεγάλο σθένος και ε, επιμονή και θα σας υποστηρίξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η κοινωνία των πολιτών. Δεν μπορεί κάθε πρόταση να παίρνει λεφτά από την αναπτυξιακή βοήθεια. Οι συνάδελφοι σας ρώτησαν πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ένα μέσο που μας απασχόλησε επανειλημμένα και πάρα πολύ για τη σταθερότητα και την ειρήνη. Τι στόχο έχει, για ποιο λόγο έχει σχεδιαστεί. Προφανώς όταν συζητάτε ε, για την ε, χρηματοδότηση λέτε ότι τα δισεκατομμύρια θα πρέπει να γίνουν τρεις εκατομμύρια. Μα πώς να το κάνουμε αυτό όταν ακόμα και οι πιο μετριοπαθείς ε, δεσμεύσεις των κρατών μελών για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια να φτάσει στο 0,7 δεν τηρούνται. και το Συμβούλιο έχει δηλώσει έτσι ξεκάθαρα ότι στην κατηγορία 4 στις νέες δημοσιονομικές προοπτικές δεν πρόκειται να αυξηθεί η πρικοδότηση. Εσείς πώς θα τα συγκεράσετε αυτά. Θα πρέπει να δούμε από κοινού πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Η νέα λοιπόν συνένεση έχει σημασία, δεν αντιλέγω, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Και τώρα τα βλέπουμε όλα αυτά να συγχωνεύονται με μια ευρύτερη διαδικασία υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων των εφόρων. Και τι είναι αυτό το κλάστερ του κυρίου Τίμερμαν τώρα που κατέβασε στην ανακοίνωση, αν κατάλαβα καλά. Είναι μια ανακοίνωση για ένα βιώσιμο μέλλον, ε, που εξετάζει και συμπεριλαμβάνει εξωτερικές και εσωτερικές προκλήσεις. Τι είναι όλα αυτά. Θα τα ανακατεύσουμε όλα μαζί, είναι κάτι διαφορετικό. Τα ρίχνουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Σίγουρα είναι πολλά ε, αυτά που μας είπατε και είναι και πολλά θετικά και συμφωνούμε με πολλά. Όταν μιλήσατε για τους βασικούς ε, ε, φορεί που μπορεί να είναι κινητήρια δύναμη, κάποιε παράμετροι όπω είναι θέματα φύλου ή θέματα επενδύσεων. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα, θα πρέπει να κυριαρχούν στη συζήτηση. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε και βέβαια πιο ισχυρέ εταιρικέ σχέσει. Επανέρχομαι όμω στη χρηματοδότηση. Οι πάντε κατανοούν ότι πραγματικά τα δισεκατομμύρια πρέπει να γίνουν τρει εκατομμύρια. πώ θα γίνει αυτό εν μέρη με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Ταυτόχρονα όμως δεν θα μπορούσατε να βεβαιωθείτε ότι ο ιδιωτικό τομέα κάπως θα πρέπει να λογοδοτεί για τον αντίκτυπο που έχουν οι επενδύσεις του στην ανάπτυξη. Αλλιώς και πάλι θα δούμε να διοχετεύονται τα χρήματα της ανάπτυξης σε αλότριους στόχους ή που δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Έχει έρθει η ώρα πιστεύω και αυτή η συζήτηση να γίνει για την εταιρική ευθύνη και λογοδοσία. Το είπε και ο συνάδελφος Λίτς. όπου συμμετέχει και ο ιδιωτικός τομέας και αναλαμβάνει και την ευθύνη του. Και ένα τελευταίο. Μιλήσατε για μια διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς. Εξ όσων γνωρίζω, η κοινωνία των πολιτών είναι απογοητευμένη γιατί δεν εισακούεται. Και πρόεδρε, μια που έχουμε και λίγο χρόνο, δεν θα μπορούσαμε να καλέσουμε κάποιον εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών έναν ή δύο να μιλήσουν γιατί αντιμετωπίζουν μια ε, πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Σε 100 περίπου χώρε συρρυκνώνεται αυτή τη στιγμή ο δημόσιο χώρο για την κοινωνία των πολιτών και εμεί θα πρέπει να την επερασπιζόμαστε και στην παρούσα διαδικασία και μετά την συνένεση. Merci, cher collègue. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε τελευταία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, συμφωνώ 100% δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Δεν υπάρχει και πολύ περιθώριο να διαφωνήσει κανείς με αυτά που είπατε. Ούτως ή άλλως αυτά που είπατε αποτελούν τμήμα του, των επιθυμιών που έχουμε εκφράσει και εμείς ε, εδώ στο Κοινοβούλιο. Να συμπληρώσω αυτά που είπαν ε, οι συνάδελφοι. Καταρχά, συμφωνώ με όλους εσάς ε, θυμάστε ότι πριν από ένα χρόνο ήμασταν στη Νέα Υόρκη ε, χαρούμενοι, γιορτάζαμε ε, μία δέσμευση που υπόγραψαν όλες οι χώρες ε, του ΟΗΕ για την ατζέντα του 2000. Ένα χρόνο μετά ξεκινάει μια ανησυχία παρόλα αυτά. Έχουμε μια αίσθηση ότι τίποτα δεν έχει κινηθεί, ούτε το πρώτο, το ένα μελιτέο βηματάκι δεν έχουμε κάνει. Είμαστε σε μια στιγμή κρίσιμη για αυτή την συνένεση ούτω ώστε να, γίνει, να εξυπηρετήσει κάτι. Είναι καλό που συμφωνούμε τουλάχιστον εμεί οι δύο Κομισιόν και Κοινοβούλιο. Αλλά είναι σαφέ ότι αν τα κράτη-μέλη, οι χώρε οι οποίε υπέγραψαν αυτή την ατζέντα, που υπέγραψαν αυτού του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη, δεν αρχίσουν την πορεία αυτή, δεν πρόκειται να φτάσουμε πουθενά. Το Συμβούλιο δεν έχει δεν εξυπηρετεί τίποτα. Όταν η κάθε χώρα που είναι ο φορέα δεν αισθάνεται ότι την αφορά αυτό το πράγμα, δεν δίνει το παράδειγμα. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει ένα μοντέλο δωρητή και ε, αποδέκτη, ας πούμε. Θα πρέπει όλες αυτές οι χώρες να υποστηρίζουν αυτούς τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Και αυτή η συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη έδειξε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να αλλάξουμε ε, το θεσμικό μοντέλο της χώρας. Και στην Ισπανία, στη χώρα μου, που είναι μια χώρα που έχει μακρά ιστορία στην αναπτυξιακή συνεργασία, πέρα από τις πολιτικές κινήσεις που γίνεται και την απουσία σταθερής κυβέρνησης, αυτή η τελευταία βουλή που προέκυψε πριν από λίγο ε, δεν είχε κοινοβουλευτική επιτροπή, ε, κοινοβουλευτική επιτροπή ανάπτυξης αυτό το κοινοβούλιο. Αλλάζει το μοντέλο. Δεν υπάρχει πια αυτή η κατακαιρμάτιση θεωρούμε τα Υπουργεία Ενέργειας, Οικονομίας, Ισότητας, Γεωργίας κτλ. θα πρέπει να έχουν και να εσωματώσουν τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλιώς δεν θα φτάσουμε πουθενά. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Σε σχέση με το ποιοι είναι οι φορεί. Μιλάμε μονίμω για την κοινωνία των πολιτών. Και μοιάζει ότι θεωρούμε ότι η κοινωνία των πολιτών ίσον ΜΚΟ. Και ότι ΜΚΟ σημαίνει μη κερδοσκοπικέ οργανώσει. Όμω, είναι σαφέ ότι και οι επιχειρήσει είναι τμήμα τη κοινωνία των πολιτών. Φυσικά η ΜΚΟ είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σωστά τα λόγια και στο διάλογο, ε, στη συμμετοχή όλοι οι φορεί τη κοινωνία θα πρέπει να συμμετάσχουν. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι οι επιχειρήσει είναι κάτι ξεχωριστό και θα πρέπει να τι αντιμετωπίσουμε με δυσπιστία και προσοχή. Όχι από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις και αυτές είναι τμήμα αυτής της συνένεσης αναγκαστικά. Θα πρέπει να αλλάξουμε αυτό το μοντέλο ε, όπου μόνο ένα τμήμα της κοινωνίας των πολιτών λαμβάνουμε μονίμως υπόψη. Επαναλαμβάνω, από τους πιο μικρούς επιχειρηματίες μέχρι τους ε, σημαντικούς επιχειρηματίες, μέχρι τις πολυεθνικές, όλοι αυτοί θα πρέπει να εμπλακούν. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, πώς, θα δημιουργήσουμε, αν θέλετε, εταιρικέ σχέσεις με τις μεγάλες επιχειρήσεις που θα επενδύσουν μετά. Θα πρέπει να αισθάνονται ε, ότι τους απασχολεί, ότι είναι δική τους αυτή η ιστορία της ανάπτυξης. Και ένα τελευταίο σχόλιο για την ε, παγκόσμια στρατηγική που δημοσίευσε η κυρία Μογκερίνη και που θα μας την διαμηνήσει προσεχώς. Το βασικό στοιχείο, νομίζω, αυτής της στρατηγικής είναι μια επιμερισμένη θεώρηση και μια κοινή δράση. Αυτά τα δύο σημαίνουν ότι αυτή η παγκόσμια στρατηγική θα πρέπει να προωθήσει τα συμφέροντα των πολιτών. Και λέει το, κείμενο ότι γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει προς την ευημερία των λαών της. Η ευημερία θα πρέπει να είναι κοινή και θα πρέπει να συνάδει με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Μια ευημερούσα Ευρώπη θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνει ένα οικονομικό ε, διεθνές σύστημα δίκαιο, ανοιχτό και μια βιώσιμη πρόσβαση στα κοινά αγαθά. Αυτό είναι προϋπόθεση. Είναι σημαντικό να έχουμε αυτή την ε, ανοιχτή θεώρηση, αυτό το ανοιχτό όραμα. Γιατί αν εμεί έχουμε αυτή την άποψη μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είμαστε όσο να είναι πολύ περιορισμένο όργανο, μπορούμε να κάνουμε λίγα πράγματα, δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Επίτροπο για να απαντήσει, να αντιδράσει στις παρεμβάσει. Έχετε το λόγο κύριε Μίμητ. Thank you very much indeed, ξεκάθαρα και να αντανακλάτε και στη συνένεση. αυτή οι σύνδεσμη αυτές οι σχέσεις, οι διασυνδέσεις, όπως θέλετε πείτε το αλληλεξάρτηση διαφόρων ε, στοιχείων της πολιτικής μας και πτυχών. Η αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί πια να είναι απομονωμένη μία συγκεκριμένη πολιτική που θα καλύπτει και θα ικανοποιεί όλες τις ανάγκες ε, του απανταχού της γης. Οπότε, η σύνδεση αναπτυξιακής βοήθειας και ε, ανθρωπιστικής, ανάπτυξης ε, και ασφάλειας, ανάπτυξη και ειρήνης ε, θα πρέπει να είναι σημαντικό στοιχείο της νέας συνένεσης. Βεβαίως, αυτό μας φέρνει ε, πολλά ερωτηματικά για τις προειδοποιήσεις, για τις ανησυχίες, για τις επικρίσεις που ακούμε σε περικές περιπτώσεις. Αλλά έχουμε ε, καλές απαντήσεις και καλά επιχειρήματα για να ε, τεκμηριώσουμε με σωστό τρόπο και το καλύτερο δυνατό αυτή τη νέα σύνδεση. Παράδειγμα, αναπτυξιακή ε, βοήθεια και ανθρωπιστική βοήθεια η συνέντευξη θα πρέπει να τονίσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μια νέα σύνδεση αυτών των δύο. Ιδιαίτερα όταν διαχειριζόμαστε τις διαρθρωτικές ε, κρίσεις, τις επίμονες που διαιωνίζονται και δημιουργούν ευαίσθητες και έφταξτες καταστάσεις. Εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη σύνδεση, ε, κοινός συντονισμός, κοινός σχεδιασμός. Ε, χρησιμοποίηση μέσων με τρόπο πραγματικά συντονισμένο. Ας πούμε στην υγεία και στην βασική εκπαίδευση. Είναι και αυτό εξίσου τμήμα και ανθρωπιστικής βοήθειας και μακροπρόθεσμα αναπτυξιακής βοήθειας. Και εκτός από τη βραχυπρόθεσμη αναπτυξιακή, μάλλον ανθρωπιστική βοήθεια και πιο μακροπρόθεσμη βοηθάει. Άρα, δεν θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας μόνο ε, ε τις ε, ανθρωπιστικές ανάγκες και την ε, σύνοδο κορυφής για τα ανθρωπιστικά θέματα. Αλλά θέλω ε, να φαίνεται αυτός ο σύνδεσμος να καθορίζεται πάρα πολύ καλά στη συνένεση για την ανάπτυξη. Υπήρξαν και προτάσεις και συζητήσεις μήπως χρειάζεται μία μόνο συνένεση για θέματα αναπτυξιακά και ε, ανθρωπιστικά. Προς το παρόν δεν έχουμε πάει τόσο μακριά να ζητήσουμε ενιαία συνένεση και για τα δύο. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά για να καλύψουμε ένα έδαφος το οποίο ε, δεν ε, είχε ακόμα χαρτογραφηθεί. Ενώ εδώ δεν είχε συνδεθεί περισσότερο με την ανθρωπιστική ε, συνεργασία. Αντίστοιχα θα μπορούσαν να λεχθούν και για την μετανάστευση και πώς αυτή συνδέεται με την ανάπτυξη. Εδώ πραγματικά χρειάζεται σύνδεση έτσι ώστε να εξυπηρετούμε τον ίδιο στόχο, διότι η μείωση της φτώχειας και η αντιμετώπιση ε, των βασικών αιτίων της ε, άτακτης μετανάστευσης και ε, της αναγκαστικής εκτόπισης είναι πράγματα αλληλένδετα. Αν δεν ρυθμίσεις το ένα δεν πρόκειται να ρυθμιστεί το άλλο. Αντιμετωπίζουμε με τη φτώχεια ε, και από την άλλη τη μειώνουμε ε, και αυτό είναι βασικό στόχος της αναπτυξιακής βοήθειας αλλά αγγίζει και τη μεταναστευτική πολιτική. Είναι λοιπόν αυτά αλληλένδετα και θα πρέπει βραχυπρόθεσμα να αυξηθούν οι ευκαιρίες που έχουν οι άνθρωποι στις χώρες τους έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Και ταυτόχρονα θα μειωθεί και η πίεση που οθεί τους ανθρώπους στη μετανάστευση γιατί φεύγουν, γιατί δεν έχουν ευκαιρίες στη χώρα τους. Ξέρω ότι μπορεί να ανησυχούν ορισμένοι με την αμυγή ε, έννοια της αναπτυξιακής πολιτικής που βασίζεται στην επίσημη κρατική βοήθεια. Αλλά αν δείτε και πάλι τα στοιχεία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν ε, χρησιμοποιηθεί από εκεί κονδύλια για άλλους στόχους, ούτε μειώθηκαν. Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, τα 68 δισεκατομμύρια, σήμαιναν αύξηση 3,6 δις ευρώ. από την ε, κλασική βοήθεια, την αναπτυξιακή, την επίσημη ODA. Ακόμα και αναφερήσετε το κόστος για τους πρόσφυγες. Λοιπόν, θέλουμε να αυξήσουμε και τα δύο και τα καταφέραμε. Την υποδοχή των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, την ανθρωπιστική αναπτυξιακή βοήθεια καλύτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε και στο μέλλον. Έρχομαι τώρα σε θέματα ασφαλείας και πώς αυτά συνδέονται με την ανάπτυξη. Και πάλι συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει μια προϋπόθεση εδώ για να επιτύχει αναπτυξιακή πολιτική. Και αυτή είναι η ειρήνη, σταθερότητα ε, στις κοινωνίες, στο περιβάλλον και στις χώρες αυτές. Προσπαθούμε λοιπόν τώρα να συνδέσουμε την ασφάλεια, την ειρήνη με την ανάπτυξη. Και θέλουμε να συμπεριλαμβάνεται και αυτό στη συνένεση με όρους πολύ σαφείς. Σε σχέση με αυτό πρέπει να σας πω ότι έχουμε δύο βασικές κόκκινες γραμμές που ποτέ δεν πρόκειται να παραβιάσουμε. Πρώτη, θα πρέπει να φροντίσουμε τα θέματα της ασφάλειας με τα, οποία μας απασχολούν ως προς την αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα φτάσουν ποτέ σε επίπεδο στήριξης κάποιων στρατιωτικών δομών ή ε, όπλα, ας πούμε, ε, ε, και στρατιωτικές δομές και δυνατότητες στις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Αυτή είναι απόλυτη κόκκινη γραμμή και στις συνθήκες και της Ένωσης ότι δεν υποστηρίζουμε τέτοια στρατιωτικά ζητήματα από την αναπτυξιακή βοήθεια με τρόπο άμεσο. Uh, uh, ε, στην παρούσα φάση. Αλλά η δεύτερη κόκκινη γραμμή που επίσης δεν θέλουμε να ε, παραβιάσουμε είναι ότι η αναπτυξιακή μας παρέμβαση για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να είναι όσο γίνεται περισσότερο, για να μην πω απολύτως, ε, προσιλωμένη και να διέπεται από ε, κριτήρια επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη σαφήνεια και για τους κανόνες ODA για ε, τον τομέα της ασφάλειας. Τώρα μπορούμε πλέον να υποστηρίζουμε αστυνομία, τομείς ασφάλειας, για τη μετώπιση του βίου εξτρεμισμού, για τον έλεγχο του ελαφρόπλισμού και τέτοια πράγματα. Αυτές ε, οι δυνατότητες ε, μάλλον οικονόμηση δυνατοτήτων, ε, οικονόμηση δυνατοτήτων για την ασφάλεια εντάσσεται στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και προβλέπεται με βασικές ασφαλιστικές δικλίδες οι οποίες είναι γνωστές και δεδομένες. Και αυτό θα τηρείται πάρα πολύ αυστηρά και θα ελέγχεται. Αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε τώρα ή αργότερα στην νομοθετική διαδικασία, γιατί είναι τμήμα αυτό για το μέσο για τη σταθερότητα και την ειρήνη. Μπορούμε να το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα της ε, νομοθεσίας για την νομική βάση, αν είναι η σωστή ή όχι. Και αν η θετική λίστα ή η αρνητική των εκτάκτων περιστάσεων και των εξαιρετικών συνθήκων είναι καλύτερη. Δεν ξέρω. Εδώ είναι ένας τομέας που πραγματικά ε, θέλουμε να συζητήσουμε στην κανονική νομοθετική διαδικασία για να καταλήξουμε στους τελικούς ορισμούς. έτσι ώστε το μέσο για την ειρήνη και την ε, σταθερότητα ε, να είναι το καταλληλότερο. To, to develop the... Έτσι ώστε να αναπτυχθεί αυτός ο σύνδεσμος ανάμεσα ε, στην ανάπτυξη και την ασφάλεια. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το εξής. Η δική μας συνένεση δεν φέρνει μόνο νέες προσεγγίσεις, η νέα πολιτική προσέγγιση ε, προς τους στόχους ε, ανάπτυξης, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να χειραφετηθούν οικονομικά οι αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε λοιπόν τρεις μεγάλες πρωτοβουλίες τουλάχιστον ε, που συνδέονται με την κοινωνική εταιρική ευθύνη ή που συνδέονται με την ενίσχυση της ε, ε, αλυσίδας παραγωγής αξίας στην εκάστοτε χώρα. Είτε πρόκειται για ξυλία, είτε πρόκειται για ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές κτλ. Τώρα υπάρχει και η πρωτοβουλία Garment, στην οποία αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως. για να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Παραλαμβάνω σε προϊόντα πώς είναι η ξυλία ή τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές. Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Η πρωτοβουλία Garment μας ε, βοηθάει να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Ε, βέβαια, ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει το στόχο. Προσπαθούμε να ε, εντάξουμε αυτή την προσπάθεια στην κλωστοεφαντοργία ως ε, βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής. Τα, βασικά στοιχεία είναι η χνηλασιμότητα, ε, αύξηση της συνειδητοποίησης των καταναλωτών, ε, υλοποίηση και επιβολή των υφισταμένων κανόνων. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το παγκόσμιο εμπόριο, που είναι σημαντικό βεβαίω να συμμετέχει και ο εμπορικό τομέα στην πρωτοβουλία αυτή για τα κλωστοφαντουργικά. Αυτό που θα θέλαμε είναι να τους επιτρέψουμε να προσθέσουν νέα αξία στην αλυσίδα παραγωγής. Ε, σε αυτό το κλάδο Τη υφαλουργία στη χώρα τους και να μην φεύγει η αξία, να μην του την αφαιρούμε από την παραγωγή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι τμήμα τη γενικότερη συνένεσης. Για την κοινωνία των πολιτών και τη συμμετοχή των ΜΚΟ συμφωνώ. Έχει σημασία να συμπεριλαμβάνουμε εκεί όχι μόνο στη δημόσια διαβούλευση, στο σχεδιασμό ε, της συνένεσης ε, να συμμετέχουν ΜΚΟ και η κοινωνία των πολιτών και οι πάντες, όχι μόνο λέγω στο στάδιο της διαβούλευσης, αλλά είναι σημαντικό στην αναπτυξιακή πολιτική να έχουμε στο πλευρό μας παραστάτη την κοινωνία των πολιτών ε, καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης πολιτικής, όχι μόνο στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή και στην υλοποίηση. Γι' αυτό η Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ ήδη αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι τον άλλο μήνα θα διοργανώσει ένα διαρθρωμένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών για τη συνένεση και για άλλα θέματα ανάπτυξης. Αυτός ο διάλογος θα γίνει μόνιμος, διαρθρωμένος δεν θα είναι άπαξ ε, για τη χάραξη της συνένεσης, θα γίνει μια μόνιμη δομή τουλάχιστον άπαξ ετησίως ε, στη διαδικασία αυτή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής και ηγέτης ε, στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ένα από τα στοιχεία που ακούσαμε ήταν ο κοινός προγραμματισμός. Βεβαίως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ως κατευθυντήρια γραμμή στη συνένεση. Ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση αυτή με τα κράτη-μέλη σε επίπεδο τεχνικών παραγόντων και εμπειρογνωμών, αλλά και σε πολιτικό, με, τις, ε, με τους Υπουργούς Αναπτυξιακής Βοήθειας. Και η συνένεση θα πρέπει να καλύπτει και τα δύο επίπεδα και το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διαχειρίζεται τα αναπτυξιακά κονδύλια αλλά και το επίπεδο ε, αναπτυξιακής βοήθειας των κρατών μελών. Και η συνέντευξη θα πρέπει να βοηθάει και να οθεί να υπάρχει ένας κοινός προγραμματισμός, σχεδιασμός και η κοινή εφαρμογή. Και αυτό να είναι ο κανόνας στη δράση μας. Είμαστε σε φάση τώρα να εγκαταλείπουμε τα εθνικά ε, ενδεικτικά προγράμματα ως μεθοδολογία ή ως εργαλείο υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων και έχουμε περάσει σε κοινό προγραμματισμό και ε, τα γνωρίζετε αυτά και ε, σε πολλά κράτη-μέλη και όσο γίνεται σε περισσότερες χώρες τέρους μας. Επίσης, θα θέλαμε να έχουμε σαφείς κατευθυντήρες γραμμές στην συνένεση για την υποστήριξη προγραμμάτων τα οποία εφαρμόζονται άμεσα ή ε, όπου συμμετέχουν οι τοπικές κοινότητες, οι τοπικές κοινωνίες και η τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο η κεντρική κυβέρνηση κάθε χώρας. Αυτό και αν είναι σημαντικό. Δίλημα. και παλιό κατά τα άλλα στην αναπτυξιακή πολιτική. Να ε, υποστηρίζουμε έργα επιτόπου με την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο με τις κεντρικές κυβερνήσεις. Έτσι πραγματικά τα έργα μας θα εκτελούνται όσο γίνεται πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες του κόσμου. Λοιπόν, πολλά μπορούμε να κάνουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή χωρίς να περνάνε όλα από βαριές κυβερνητικές διαδικασίες και αποφάσεις μέχρι να φτάσουν στον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Έτσι, αυτό κάπως πρέπει να το δούμε. Δεν θέλει κανείς να, να παρακάμψει, να βραχικυκλώσει την κυβέρνηση, αλλά να, να έχουμε προγράμματα και σε συνεργασία άμεση με την τοπική κοινωνία και να συνεχίσουμε να πιέζουμε τις κυβερνήσεις. Αλλιώς η δράση μας δεν πρόκειται ποτέ να πιάσει τόπο, ούτε οι λύσεις να είναι ε, μόνιμες και βιώσιμες, ούτε οι κυβερνήσεις καλύτερα. Αν εξακολουθήσουμε την παλιά αναπτυξιακή συνεργασία σε επίπεδο κυβερνήσεων. Αυτά. Τελειώνοντας. Πραγματικά προσβλέπω στη συζήτηση που θα έχουμε για να συνεργαστούμε για τη συνένεση έτσι ώστε να γίνει μια μόνιμη συνεργασία με τους παλιούς τους γνωστούς εταίρους, ε, τα τρία θεσμικά όργανα, αλλά και την κοινωνία των πολιτών και άλλους φορείς. Διότι είναι ο μόνος τρόπος αυτός για να μπορέσουμε να μεταφράσουμε αυτό το νέο στοιχείο που είναι και επαναστατικό η ε, στόχη της βιώσιμης ανάπτυξης να μεταφραστεί λίγο στην πράξη, στην πραγματική ζωή. Ευχαριστώ και πάλι για τις ιδέες σας, για τις προτάσεις σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κοινή δουλειά που μας περιμένει έτσι ώστε να φέρουμε τη συνένεση σε αίσιο πέρας. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Κύριε Χάουτα, θα να ξαναπάρει το λόγο. Σύντομα. Ο κύριος Γκέρεντς θέλει να ξαναπάρει το λόγο. <coughs> Ε, Ευχαριστώ, Να συμφωνήσω με την κυρία Χάουταλα. Πρέπει να οργανώσουμε μια συνέχεια σε αυτήν εδώ τη συνεδρίαση. Κάναμε, κάναμε μια καλή ανταλλαγή απόψεων. Θα πρέπει όμως να εμπλέξουμε και όλους τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς και να γίνει και λίγο πιο αμφίδρομη δεν ξέρω αν συνεχίζει το διαθέμενο διάλογο η Κομισιόν με εκπροσώπους των κρατών μελών. Ναι, ναι, γνέφει η Κομισιόν. Να σας κάνω μια υπόδειξη, αν μου επιτρέπετε. Καλό θα ήταν να συζητήσει ο διαθέμενος διάλογος αυτό το θέμα. Αυτό ζητάω. Επίσης θα πρέπει να οργανωθούμε εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Γιατί και τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να πούν δύο λόγια. Εκείνοι ψηφίζουν του προπολογισμού, εκείνοι προωθούν τι πολιτικέ σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε να κάνουμε πολλά λοιπόν. Μωρή, σε εμπιστεύομαι για να στείλει αυτό το μήνυμα στο Προεδρείο τη Επιτροπή μα για να οργανωθούν όλα αυτά. Τι προθεσμία έχετε, Ποιε είναι οι επόμενε εκδηλώσει, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Περιμένουμε τη συνέχεια, Μωρίς. Σύντομα. Δίνω το λόγο στον κύριο Για τους ΜΚΟ. Δεν είναι σωστό στην, στο τέλος της συνεδρίαση να λέμε ότι κάποιος από τις ΜΚΟ θα πρέπει να έρθει και να σχολιάσει τον επόμενο μήνα θα εμπλακούν οι ΜΚΟ σε μια ειδική συνεδρίαση. Και είναι πολύ καλό αυτό να ακούσουμε τις ιδέες και τις προτάσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών θα πρέπει να μιλήσουμε για τη σημερινή συνεδρίαση και τις συνέπειες που απορρέουν από αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο ξανά στον Επίτροπο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 ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε την έκθεση της Επιτροπής μας και νομίζω ότι και αυτή η έκθεση θα συνεισφέρει για να δημιουργηθεί η νέα συνένεση. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, έχουμε το σημείο 4 και με αυτό θα τελειώσουμε. Θέλει να πάει κανένα τώρα στα διάφορα. Ουδής. Σημείο 5. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου του 2016 από τις 8.30 μέχρι τις 10 στο Στρασβούργο. Θα παρουσιάσουμε το θέμα του βραβείου, του υποψήφιου δηλαδή για το βραβείο Σαχάροφ. 10 Οκτωβρίου του 2016 από τις 3 μέχρι τις 6 ε, στις Βρυξέλλες και από τις 9 μέχρι τις 12.30 και από τις 3 μέχρι τις 6.30 στις 11 Νοεμβρίου. Τελειώνει εδώ η συνεδρίασή μας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας.